φέροντα των φορολογούμενων ε, και να αποκομίσουν θετικά ωφέλη οι κάτοικοι αυτών των περιοχών. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι. Το επόμενο και τελευταίο σημείο στη μίση διάταξη είναι η έκθεση της συναδέλφου κυρίας Γκρέζ με θέμα αναπτυξιακές πτυχές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε θέματα γενετικών πόρων. Δίνω το λόγο στην ε, εισηγήτρια για τέσσερα λεπτά. Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Μετά από μια μεγάλη και μακρά διαδικασία, την 6η Δεκεμβρίου του 2012, η έκθεση ε, για τις ε, ε, επιπτώσεις των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τους γενικού πόρους ε, για τις αναπτυσσόμενες χώρες και τις επιπτώσεις της μείωση της φτώχειας εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Είναι μια σημαντική μέρα αυτή της υπερψήφισης γιατί για πρώτη φορά Ευρωπαϊ, Ευρωπαίοι βουλευτές από όλα τα πολιτικά κόμματα και όλους τους σχηματισμούς συμφώνησαν ότι θα πρέπει να σταματήσει η λαϊλεσία των γενετικών πόρων στον πλανήτη μας. Δεν είναι πλέον ταμπού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η λέξη βιοπειρατεία και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως όλους τους συνδέλφους που συμμετείχαν σε αυτήν την σημαντική διαδικασία. Αύριο θα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο όμως. Η ψηφοφορία είναι σημαντική έτσι ώστε να ε, εκφράσουμε την αποφασιστικότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο σύνολό του να προχωρήσει έτσι ώστε οι πολιτικές ανάπτυξης να αποκτήσουν μεγαλύτερη συνεκτικότητα. Θα πρέπει να επανατοποθετηθούμε ε, ε, απέναντι στην βιοπειρατεία, να ε, δεσμευτούμε στην υπεράσπιση των τοπικών οικονομιών, των παραδοσιακών γνώσεων, του σεβασμού, των δικαιωμάτων, των αυτοχθόνων και των μικρών καλλιεργητών. Και τέλος να δεσμευτούμε ότι θέλουμε να διατηρήσουμε το περιβάλλον και την βιοπικιλότητά του. Γνωρίζετε ότι 90% του βιολογικού, ε, της βιολογικής παγκόσμιας κληρονομιάς βρίσκεται στις αναπτυσσόμενες χώρες. Όμως ε, ε, η μεγαλύτερη πλειοψηφία των ε, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ανήκουν στις αναπτυγμένες χώρες. Γνωρίζουμε ότι οι γενετικοί πόροι έχουν τεράστια σημασία για την αηφόρο γεωργία και την διατροφική ασφάλεια σε ολόκληρο τον κόσμο προστασία λοιπόν της ε, ε, ε, γενετικής ποικιλία, διατήρηση της ιδείας. Αυτές είναι οι λέξεις κλειδιά έτσι ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι της χιλιετίας για την ανάπτυξη. Πρέπει να επαναφερθούμε στην αρχή της ορθής ανάπτυξης και έτσι όπως αναφέρεται στο άρθρο 208 της Συνθήκης της Λισαβόνας οι κανόνες που συνοδεύουν αυτή τη ε, ε, στιγμή την εκμετάλλευση των ε, πόρων και των παραδοσιακών γνώσεων καθορίζονται ελιπέστατα. Επομένως, αυτό το νομικό κενό δίνει την δυνατότητα σε κάποιες μεγάλες εταιρείες να επωφεληθούν έτσι ώστε να λαιλατίσουν αυτό το παραδοσιακό κεφάλαιο γνώσης επίσης ε, αυτά τα θέματα τα διαχειρίζονται ε, πάρα πολλές κατακαιρματισμένες οργανώσεις ε, και αυτό βοηθάει περισσότερο όσους θέλουν να βρουν το δρόμο τους ανάμεσα σε, αυτούς, τους, σε αυτά τα κενά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε υπογράψει το πρωτόκολλο της Ναγκόγια και θα πρέπει να το υλοποιήσουμε. Θα πρέπει να αναλάβουμε τις ε, ε, ευθύνες μας ε, και να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες στις προσπάθειές τους βάσει των οποίων θα πρέπει να ζητηθεί άδεια από τις αναπτυσσόμενες χώρες να υπάρχει ρητή συμφωνία τους και τέλος να μοιραστούν τα ωφέλη. Θα πρέπει να καταδικάσουμε ρητά κάθε πρακτική η οποία αντιτίθεται στις δεσμεύσεις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει όσον αφορά τη διατήρηση της βιοπικιλότητας. Ε, στηρίζομαι πάνω σας για το αποτέλεσμα της ευρωενής ψηφοφορίας και σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Ναι, κυρία Ισηγήτρια, διαδικασία Catch the Eye. Δίνω το λόγο στον συνάδελφο κύριο Πάσκα. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda komisie. Počas Γνωρίζουμε ότι κάποια φυτά τα οποία καλλιεργούνται από τοπικές κοινότητες στον κόσμο και οι παραδοσιακές γνώσεις για την δράση των συστατικών του ουσιών χρησιμοποιούνται από μεγάλες βιομηχανικές και φαρμακευτικές χημικές επιχειρήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και κατοχυρώνονται στο όνομά τους οι πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται από, τις, από τους ηθαγενείς ε, πληθυσμούς δυστυχώς ε, γίνονται αντικείμενο κατάχρησης και προστασίας από τους λεγόμενους βιοπειρατές, βιολογικούς πειρατές. Και οι πραγματικοί δημιουργοί δεν έχουν κανένα όφελος από τη βιομηχανική χρήση των ουσιών αυτών. Πρέπει να τροπολογήσουμε τη συμφωνία TRIPS έτσι ώστε να είναι συμφατή με το πρωτόκολλο της Ναγκόγια. Μόνο με τον τρόπο αυτό θα αποτρέψουμε την κατάχρηση των παραδοσιακών γενετικών πόρων και γνώσεων. το λόγο στη συνάδελφο κυρία Αντρές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για τη συνένεση που έλαβε από όλε τι ε, πολιτικέ ομάδε. Καταρχήν είναι προφανές ότι οι φυσικοί πόροι από τα φάρμακα μέχρι τα καλλιτικά προέρχονται από αναπτυσσόμενες χώρε. Αλλά τα ωφέλη είναι για τι επιχειρήσει και τα εργαστήρια, όχι για αυτέ τι ε, ε, κοινότητε που τι παράγουν. Ε, η έκθεση ομιλεί για τη δυνατότητα τα πράγματα να αλλάξουν και τα ωφέλη ε, να προορίζονται και στις ε, χώρες αυτές που παράγουν τους σπόρους. Έχουμε καταθέσει κάποιες θεωρολογίες όσον αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας καθώς και την υποχρέωση δημοσιοποίησης της πηγής προέλευσης των γενετικών πόρων ούτω ώστε να αποφελούνται οι τοπικές κοινότητες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει τη συνένεση μετά από την ενημέρωση των κοινοτήτων. Ε, υπάρχει ο κίνδυνος απαγόρευσης κάποιων παραδοσιακών σπόρων. Ε, θα πρέπει να να, νομίζω θα πρέπει να υποστηρίξουμε την επιστημονική έρευνα και με τον τρόπο αυτό θα υποφεληθούμε όλοι μας. Κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει πράγματι να προστατεύσουμε τη βιοπικιλότητα. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση των πιέσεων που υφίσταται το περιβάλλον σήμερα. Η προστασία επίσης της βιοπικιλότητας και της ποικιλότητας της γενετικής είναι ε, κάτι το απαραίτητο. Τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας πάνω στις παραδοσιακές γνώσεις των χωρών ιδιαίτερα από υπό ανάπτυξη είναι απαραίτητο να προστατευθούν η γενετική πόρη είναι απαραίτητη επίσης για να υπάρξει στο μέλλον μια αηφόρος γεωργία και να διασφαλιστεί η προμήθεια τροφίμων για τον πληθυσμό της γης. Θα πρέπει οι διαδικασίες προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας να είναι συμβατές με ε, την ανάπτυξη και με τον σεβασμό για το περιβάλλον. Ε, στο σύμφωνο της Ναγκόγια είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να υπογραφεί το ταχύτερο δυνατόν και να διασφαλιστεί η δικαιοσύνη. Κύριος Φερέιρα. Ζωάου Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σε ένα πλαίσιο μιας ε, παγκόσμιας αλλαγής, ο γενετικός παράγων είναι παράγων ε, κλειδί για τα οικοσυστήματα. Τα, ε, η διαφοροποίηση των διαφόρων φυτικών ειδών είναι πολύ σημαντική όσον αφορά τη διατροφή αλλά και τα πνευματικά δικαιώματα είναι εξαιρετικά καθοριστικά. Άρα θα πρέπει να υπάρξει μια συνολική αξιολόγηση. Η γενετική ε, πόρη της γης είναι κοινό αγαθό και διαφύλαξή τους θα πρέπει να γίνει από κοινού. Ε, καμία χώρα δεν θα πρέπει να αποκλείεται από τις επιστημονικές ε, εξελίξεις που βασίζονται ακριβώς στη βιοπικιλότητα των γενετικών πόρων στο διαδροφικό τομέα, στον τομέα της υγείας τα φάρμακα ε, ε, την παραγωγή των φαρμάκων ε, πολλοί αποκλείονται από όλες τις διαδικασίες και αυτό είναι μια απόδειξη εξέλιξης του καπιταλισμού. Εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κυρίως την κυρία Γκρέζ για την έκθεση της για τις αναπτυξιακές πλευρές της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Ευχαριστώ τις επιτροπές που ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο για να υπάρξει σωστός έλεγχος των διαδικασιών αυτών. Όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, θα βοηθήσει η προστασία αυτή να καταπολεμηθεί η πείνα στον κόσμο. Θα προωθηθεί η έρευνα, η επιστήμη, και ε, θα αποδειχθεί ακόμα περισσότερο το εμπορικό και οικονομικό ενδιαφέρον της βιοπικιλότητας. Η βιοτεχνολογία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και μπορεί να καταπολεμήσει επίσης και τη φτώχεια. Είδαμε όμως ότι υπάρχουν αυξημένες ανησυχίες από τις αναπτυσσόμενες χώρες για την κατάχρηση των γενετικών του πόρων και για τον τρόπο, ε, θα έλεγα, με τον οποίο δημιουργούνται κέρδη ε, μέσω ακριβώς ε, της βιοπικιλότητας για τις μεγάλες επιχειρήσεις και τις μεγάλες χώρες. Αναγνωρίζουμε τις ανησυχίες ε, των αναπτυσσομένων χωρών και προσπαθούμε να υπάρξει συνέργεια ανάμεσα στη σύμβαση την οποία προωθούμε και σε άλλες συμφωνίες σε διεθνές επίπεδο για την πνευματική ιδιοκτησία και την προστασία της βιοπικιλότητας για την παραγωγή τροφίμων. Η νέα συνθήκη και το πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την δίκαιη πρόσβαση και ισόρροπη πρόσβαση στην βιοπικιλότητα είναι νομίζω τα πεδία μέσω των οποίων θα δημιουργηθεί ασφάλεια για όσους θα ήθελαν να εμπλακούν και να ασχοληθούν με τους τομείς αυτούς. Έτσι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε την διατήρηση της βιοποικιλότητας στις χώρες πηγές θα έλεγα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη προτείνει νομοθετικά μέτρα για την επικύρωση του πρωτοκόλου της Ναγκόγια από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το οποίο θα δώσει νομική βεβαιότητα στους ε, εμπλεκομένους από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους γενετικούς πόρους. Ταυτόχρονα η προτινόμενη ε, νομοθεσία θα επιτρέψει επίσης να ικανοποιηθούν και οι νομικές απαιτήσεις χωρών οι οποίες παρέχουν τους πόρους αυτούς. Αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά το σύνολο των αναπτυσσομένων χωρών το σύστημα αυτό δεν θα πρέπει να έχει πάρα πολύ υψηλά διοικητικά και οικονομικά βάρη για τις επιχειρήσεις, τα εργαστήρια και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Προσπαθούμε να καταλήξουμε στους μηχανισμούς που απαιτείται για την θέση σε ισχύ του πρωτοκόλου της Ναγκόγια. Υποστηρίζουμε σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή την δημιουργία ενός μηχανισμού clearing ε, σε στενή συνεργασία με άλλες περιφέρειες και χώρες έτσι ώστε να εφαρμοστούν σωστά οι συστάσεις ε, ε, του πρωτοκόλου της Ναγκόγια. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη υποστηρίζουν τις υπόλοιπες χώρες να επικυρώσουν το πρωτόκολλο. Ένα σημαντικό Παράδειγμα είναι η πρωτοβουλία ανάπτυξης πολλαπλών δυνατοτήτων από πλευράς των χωρών ΑΚΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι το μέσο αυτό είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία θα και στην οποία συνεισφέρει με σημαντικό τρόπο. Συμπληρωματικά υπάρχουν και άλλα νομικά μέσα τα οποία θα πρέπει να αναπτυχθούν. Έχουμε εμπλακεί σε συζητήσεις με τον ΠΟΕ Έχουμε προχωρήσει σε διμερείς συμφωνίες και σχέσεις με συγκεκριμένες χώρες έτσι ώστε να υπάρξει μια ισόρροπη λύση για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και να αποφευχθούν αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον, <clears throat> ε, για τη γεωργία και για την καταπολέμηση της ένδυας. Οι προτάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ένα συνεκτικό και εύκολα διακυβερνήσιμο σύστημα είναι μια λύση για τις φτωχότερε χώρε. Πιστεύουμε ότι ένα σύστημα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας το οποίο προωθεί την καινοτομία ε, και την κυκλοφορία της τεχνολογίας προς όφελος όλων και παροχαίων γενετικών πόρων ε, και ε, γενικότερα χρηστών γενετικών πόρων και παραδοσιακών γνώσεων. Πρέπει να προωθήσουμε λοιπόν τη συνεργασία με το Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα με την Επιτροπή για την Ανάπτυξη του Κοινοβουλίου. Κομισιόν, ε, τον κύριο Σεύκοβιτς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση ολοκληρώθηκε. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο το μεσημέρι στις 12. Καλή σας νύχτα.